Ποιος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 ταυτόχρονα θα κάνουμε και Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Να σας δώσω τα αποτελέσματα της πρώτης σημερινής ψηφοφορίας. Εξεταστική Επιτροπή για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά τη μεταφορά ζώων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμόρφωση αρμοδιοτήτων και σύνθεση της. Εγκρίνεται. Μετά τεχνική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, παράταση προθεσμιών, COVID, τροπολογίες 1 και 6 απορρίπτονται, 2, 3, 4 και 5 δεκτές. Μετά, ειδικέ ε, ρυθμίσεις ε, στο πλαίσιο του ELA, στο πλαίσιο του COVID-19, τροπολογία 1 δεκτή με τα προσωρινά μέτρα που αφορούν τις ε, προθεσμίες ε, για την ε, τροπολογία πολιτών για το COVID. Τροπολογίες 7, 8, 10 και 11 εγκρίνονται. Τροπολογίες 1, 2, 3 και 4 καταπίπτουν. 6, 9, 12, 13 και 14 δεκτές. Τροπολογία 5 απορρίπτεται. Μετά έχουμε μια πρώτη σειρά τροπολογιών ε, επί του ψηφίσματος που αφορά τις δηλώσεις για τον ρατσισμό Τροπολογία 30 απορρίπτεται. Παράγραψα ένα αρχικό κείμενο δεκτή, δύο αρχικό κείμενο δεκτή, τρία αρχικό κείμενο δεκτή, τέσσερα 61 ε, απορρίπτεται, τροπολογία 20 απορρίπτεται, 35 απορρίπτεται, 21 απορρίπτεται, 31 απορρίπτεται, 62 δεκτή, 5 αρχικό κείμενο και τα 3 μέρη καταπίπτουν, 22 δεκτή, 53 δεκτή, παράγραφος 6 αρχικό κείμενα σε δύο μέρη εγκρίνεται, 36 απορρίπτεται, 9 αρχικό κείμενο δεκτά και τα δύο μέρη, παράγραφος 10 αρχικό κείμενο δεκτή, τροπολογία 32 απορρίπτεται, τροπολογία 1 απορρίπτεται, 66 δεκτή, 23 απορρίπτεται, 24 απορρίπτεται, 25 απορρίπτεται, 40 δεκτή, 44 δεκτή, 67 απορρίπτεται, 14 αρχικό κείμενο καταπίπτει, 63 απορρίπτεται, 15 αρχικό κείμενο δεκτή, Τροπολογία 10 δεκτή, τροπολογία 11 δεκτή, 16 αρχικό κείμενο 2 μέρη δεκτή, 37 δεκτή, 55 απορρίπτεται, 12 δεκτή, 19 αρχικό κείμενο σε 2 μέρη δεκτή, 33 απορρίπτεται, 21 και στα 4 μέρη δεκτή, 6 απορρίπτεται, 38 απορρίπτεται, 39 απορρίπτεται, 64 απορρίπτεται, 27 απορρίπτεται, 41 δεκτή, 45 δεκτή, 65 απορρίπτεται, 13 απορρίπτεται, 46 δεκτή, 7 δεκτή, 8 απορρίπτεται, 28 απορρίπτεται, 29 απορρίπτεται, 54 δεκτή, 47 απορρίπτεται, 48 απορρίπτεται, 49 απορρίπτεται, 50 δεκτή, 2 απορρίπτεται, 14 απορρίπτεται, εκτιμώντας ε αρχικό κείμενο δεκτό, εκτιμώντας f απορρίπτεται, Τροπολογία 57 απορρίπτεται, 15 απορρίπτεται, 51 δεκτή και η τροπολογία 52 γίνεται δεκτή. Αυτά για τα αποτελέσματα της ε, ψηφοφορίας. Τα όσα δεν διάβασα μπορείτε να τα διαβάσετε και στη σελίδα του Κοινοβουλίου και περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ψηφοφοριών. Είναι 13 και 35 οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να ψηφίζουμε μέχρι τις 3 η ώρα. Έχουμε την ίδια διαδικασία ψηφοφοριών όπως και στον προηγούμενο γύρο. Άρχεται η ψηφοφορία, μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι τις 3. Ε, τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου θα γίνουν γνωστά στις 17 και 30. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.